σημείο ε, Μοχάμετ Ραμαντάν ε, η, στο Μπαχρέιν. Αρχίζουμε με τους ομιλητές που είναι και συντάκτης ε, του σχέδιου ψηφίσματος. Σμίτ, δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει καλή συνεργασία εντός εθούσης για αυτό το πάρα πολύ καλό ψήφισμα και ειλικρινά το ελπίζω όταν μιλάμε για την ε, θανατική ποινή. Υπάρχουν αυτοί στον Μπαχρέιν που θεωρούν ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με το βασίλειο αυτό και υπάρχουν και άλλες χώρες στην περιοχή και γιατί ασχολούμαστε συνέχεια μαζί τους. Μα ασχολούμαστε και με τις γειτονικές ε, χώρες και ε, δεύτερον κατά μία ανάποψη είναι γιατί έχουμε προσδοκίες από τον Μπαχρέιν. Θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει μία πρόοδος στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και μπορούν να γίνουν χρήσιμες ε, συζητήσεις. Και βεβαίω βλέπουμε μεταρρυθμίσεις προς μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ένα συνήγορο του πολίτη, Επιτροπή Δικαιωμάτων Φυλακισμένων, ειδική ομάδα έρευνών, θετικές εξελίξεις, αλλά η πρόοδος αυτή έχει καθυστερήσει και πρέπει να συνεχιστεί. Και μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη ε, διαδικασία με το να ασκούμε βεβαίω μεγαλοφωνή κριτική, αλλά και επικοδομητική κριτική και βεβαίως για την καταδίκη του κυρίου Ραμαντάν εις ε, θάνατον μαζί με εννέα άλλους ε, υπηκόους ε, του βασιλείου. Επίσης στην παράγραφο 3 τονίζουμε την ανάγκη να προστατευθούν οι υπερασίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μπορούν να δουλεύουν χωρίς παρενόχληση ο εσωτερικό διάλογος εντό ε, του Μπαχρέιν έχει μεγάλη σημασία για να ολοκληρωθεί η πρόοδο και ελπίζω λοιπόν να στηρίξουμε αυτό το ψήφισμα σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κοράο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να μην δούμε την αποτυχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση του Μπαχρέιν. Τι έχει γίνει πρακτικά, ποια θα επόμενα βήματα όταν οι ακτιβιστές παραμένουν φυλακισμένοι και έχουν βασανιστεί ή κακοποιηθεί. Έχουμε μέχρι τώρα ε, μια ε, υπέροχη ε, απουσία της συνεργασίας της εγκαλικής μεταξύ των κρατών μελών για να προσαρμοστούν οι σχέσει μα με το Μπαχρέιν και παρόλα αυτά δεν έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε του ακτιβιστέ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε τι παραβιάσει υπάρχουν σε χώρε που καταπιέζουν την ε, ε, περίπτωση τη ειρηνική διαδήλωση και τη ελεύθερη έκφραση. Οι περιπτώσει του Χουσαίνα Λιμόζα και του ε, Μοχάμεντ Ραμαντάν που ε, συνελήφθησαν με ψευδείς κατηγορίες είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτήσουμε όλα τα κατημέλη μια βασική στρατηγική για την προστασία των αλλοδαπών που κατοικούν στον Παχρέν για να μην υπάρχει οικονομική και να ασκηθεί οικονομική και διπλωματική πίεση για να απελευθερωθούν οι φυλακισμένοι που με ψεύδεις κατηγορίες έχουν βρεθεί σε κάθριξη. Ευχαριστούμε κύριο Παντζέρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ η δραματική αντιπαράθεση που φέρνει αντιμέτωπες στις χώρες του κόλπου δεν θα λυθεί εφόσον το Ιράν και η Σαουδική Αραβία προσπαθούν να επιβάλλουν την ηγεμονία του στο Μπαχρέιν. Οι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν είναι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε πολιτική αντίρρηση. Ο Μοχάμετ Ραμαντάν, με τον οποίο ασχολούμαστε σήμερα, είναι ο πολλωστό ακτιβιστή που έχει εργαστεί στο Μπαχρέιν και έχει καταδικάσει τι κυβερνητικέ πολιτικέ, ε, οι οποίε καταστέλουν τελείω τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η άλλη περίπτωση για την οποία συζητούμε, αυτή άλλων ακτιβιστών, ε, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να αφήσουν τη χώρα, συγκεκριμένα του Αμπτουλά Αλκαλίθα, ε, είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπως και η άσκηση βασανιστήριων από την πλευρά της αστυνομίας, των αστυνομικών δυνάμεων. Όλα αυτά δείχνουν τη λογική που επικρατεί για την περιορισμό της ελευθερίας της δημοκρατικής κοινωνίας και τον, την επιβολή ελέγχου στην έκφραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρόκειται για μια ιονή κατοχή και θα θέλαμε οι αρχές του Μπαχρέν επιτέλους να απαντήσουν στις δικέ μας μας για πάυση αυτών των δράσεων. Ευχαριστούμε ο κύριος Σντόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να πω ότι το ψήφισμα αυτό είναι μια τεράστια, ένας τεράστιος συμβιβασμός. Ε, συμβιβασμός από όλες τις πλευρές. Το ΕΛΚ επιτέλους στηρίζει αυτή τη συμβαστική λύση, όμως θα πρέπει να τονίσω ότι είχαμε πολλές επιφυλάξεις ως προς το κείμενο αυτό και αρχικά δεν είμαστε σύμφωνοι για την διατύπωση του κειμένου. Το κείμενο επίσης μας δείχνει κάτι ακόμα, πόσο σημαντικό είναι να επαληθεύουμε και να εξακριβώνουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Πολλές ομάδες εδώ προσπάθησαν να συμπεριλάβουν πληροφορίες στο ψήφισμα, οι οποίες δεν είναι αναγκαστικά αληθείς. Ήταν λοιπόν αδύνατον οι πληροφορίες αυτές να εξακριβωθούν βάσει των πηγών μας. Πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό θα πρέπει να εκλειφθεί ως έκκληση προς τις αρχές του Μπαχρέιν για να διερευνήσουν την περίπτωση του ε, Μοχάμεντ Ραμαντάν και όλων των άλλων ακτιβιστών που έχουν ε, κατηγορηθεί για παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κύριο Στάνο και ένα λεπτό. Υπάρχουν σαφώς θεμητές ανησυχίες όσον αφορά την σύλληψη και την δίκη του Μοχάμετ ε, Ραμαντάν και εμείς ζητάμε από τις αρχές ε, και τον ε, ΣΕΙΧΙ να διεξάγουν μια έρευνα όσον αφορά τις κατηγορίες για βασανιστήρια και να αναθεωρηθούν πιθανώς οι καταδίκες εάν αυτό απαιτείται. Όμως το προτινόμενο κοινό κείμενο θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ έντονο καταδικάζεται συνολικά αυτό το μικρό νησιωτικό κράτος που καταβάλει τεράστιες προσπάθειες ε, για να βελτιώσει την διακυβέρνηση και δεν μπορούμε άρα να το στηρίξουμε και δεν λαμβάνει υπόψη το ότι το Μπαχρέιν αντιμετωπίζει και παρεμβάσεις από το Ιράν. Η χώρα μου έχει ισχυρούς δεσμούς με το Μπαχρέιν από την ίδρυσή του ήδη, καθώς ήταν η αρχική προστάτηδα δύναμη και σήμερα βεβαίως ε, αποτελεί και ναύσταθμο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού. Κάτι το οποίο μας ε, υπενθυμίζει τους στενούς δεσμούς που έχουμε και τη σημασία του Μπαχρέιν αλλά βεβαίως και το γεγονός ότι πολλές ομολογίες γίνονται ανοιχτές στην χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Merci. Το 2011 πάνω από το μισό του πληθυσμού στο Μπαχρέν κατέβηκε σε συλλαλητήριο. Ήταν οι ΣΥΙΤΕΣ καταπιεσμένη μειονότητα, ήταν όμως δημοκρατική αντίστασή τους. Δεν είχε καμία επιτυχία γιατί η Σουηδική για τους κατέστηλε αυτή την ε, συγκέντρωση. Ε, είναι στη δεύτερη θέση το Μπαχρέν σε σχέση με τις φυλακίες και τις παράνομες κρατήσεις. Παραβιάζονται οι βασικές θεμελιώδεις ευκαιρίες και χρησιμοποιείται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και πολιτικές μεθοδεύσεις. Θανατική ποινή 10 ε, απαγγέλθηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα και ε, πάνω από 208 έχασαν την υποκότητά του τελευταίους μήνες. μήνε. οι αρχέ του Μπαχρέν θέλουν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσει. Υπάρχουν τα 26 συστάσεις από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνώμων να πρέπει να σταματήσουν τα βασανιστήρια ε, και οι ομολογίες που αποσπούν από του κρατούμενου. Μόνο με τα περιστατικά που μπορούμε να αποδείξουμε με την καλή θέληση και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι με αυτά που κάνει τον Μπαχρέν το αντίθετο αποδείκνει. Ευχαριστούμε. Σάκε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, ε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Έχουμε ακούσει επανειλημμένως από τις αρχές ε, του Μπαχρέιν ότι θέλουν να επικεντρωθούν στην ενέργεια, την ασφάλεια και άλλα θέματα ε, αμοιβαίου ενδιαφέροντό Το ακούσαμε και την τελευταία εβδομάδα. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε ξανά από τις αρχές του Μπαχρέιν να πάψουν τα βασανιστήρια, να καταπιέζουν την έκφραση τη άποψη των μειονοτήτων και να καταπιέζουν τους πολίτε και επιτέλους να σταματήσουν και την άσκηση της θανατικής ποινής. Ο Μουχάμετ Ραμαντάν είναι ένας από τους δεκάδες που περιμένουν να θανατωθούν στο Μπαχρέιν, όμως είναι ο πρώτος ο οποίος έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα. Θα πρέπει λοιπόν οι αρχές του Μπαχρέιν, τις οποίες καλούμε έντονα να ε, πάυσουν την άσκηση της θανατικής ποινής, επιτέλους να το πράξουν. Και γενικότερα ο καλύτερος και ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια υποφελή και ε, βαθιά συνεργασία μεταξύ αρχών του Μπαχρέν και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιτέλους ε, αναντήρητα να σεβαστούν τα δικαιώματα όλων των πολιτών της χώρας. Για να μπορέσει η ειδική εκπρόσωπος του ΟΗΕ να έχει πρόσβαση στη χώρα και να επισκεφθεί τα σοφρονιστικά ιδρύματα, εκεί που κρατούνται οι αντιφρονούντε, είναι απαραίτητο για να δούμε ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη. Ευχαριστούμε. Μανέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι κατά τη ε, θανατική ποινή ε, και των ε, βασανιστήριων. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για βασανιστήρια και θανατική ποινή και ελπίζω η κυβέρνηση του Μπαχρέιν να επανεξετάσει τα μέτρα αυτά. Νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν γιατί μας έχουν δείξει ότι είναι συνεννοήσιμοι όμως θεωρώ πως ε, τα ψηφίσματα αυτά όσα ψηφίσματα και να περάσουμε εμείς εδώ πέρα κατά μικρών κρατών στον Περσικό κόλπο. Όταν ε, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά θα αποτύχουν. Η Διεθνής ε, Αμνηστία μας λέει πως ε, το Ιράν είναι μία από τις χώρες εκείνες που χρησιμοποιούν την θανατική ποινή περισσότερο. Δύο-τρεις εκτελέσεις την ημέρα. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε τόσο επιλεκτικοί λοιπόν. Τα ίδια για όλους. Μόνο έτσι θα μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε και στο Ιράν. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες για ένα λεπτό. Πέντε χρόνια μετά από τις ειρηνικές διαδηλώσεις ε, στο Μπαχρέν ε, βλέπουμε έντονη ε, καταπίεση, εξαφανείς απαγωγές, βασανιστήρια, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποινές κατά των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράνομες φυλακίσεις. Χρησιμοποιείται ο τρομοκρατικός νόμος κατά των αντιφρονούντων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των κατασταλτικών καθεστώτων πρώτον. Όμως μας ανησυχεί μια, ένα νομοθέτημα που χρησιμοποιήθηκε ε, συγκεκριμένα για τη θανατική ποινή για να το επιβληθεί η θανατική ποινή του ε, Μοχάμετ Ραμαντάν μετά από βασανιστήρια ε, και αυτό θα πρέπει να είναι ένα πρώτο βήμα που θα γίνει για την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Βαχρέιν. Θα πρέπει να μετατραπεί η ποινή που επιβλήθηκε στο Μοχάμετ Ραμαντάν και επίσης θα πρέπει να ακουστεί και η φωνή των γειτονικών χωρών. Θα πρέπει να επιτραπούν οι επισκέψεις και να υπάρξει πρόσβαση σε όλους τους χώρους κράτησης. Ε, φυσικά ε, θα πρέπει να εκφράσουμε και την ελληνική μας για όλους τους κρατουμένους Ιμπραήμ Σαρίφ, Αμπτουλά Αλκαγουάτζα, Μοχάμετ Αλμουντά, Ιουσέκ Αλμισαλμάν. Τους γνωρίζω προσωπικά. Thank you. Mr. Kelly. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για το θέμα αυτό, όπως ε, και οι άλλοι συνάδελφοι. Θα ήθελα να πω πως έχει σημειωθεί σοβαρή πρόοδος από το Μπαχρέιν, το οποίο συνεργάζεται μαζί μας στον τομέα του εμπορίου και σε άλλους τομείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γνωρούμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν ε, όταν παραβιάζουν διεθνείς συμβάσεις να τους ασκήσουμε πίεση, ειδικά στην περίπτωση του Μουχάμεντ Ραμαντάν και ειδικά ε, το πώς κατέληξε η υπόθεσή του στην ε, θανατική ποινή είναι κάτι το τελείως άδικο και είναι θύμα. Πρέπει να συσταθεί μια ομάδα εργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μπαχρέιν για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ward, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη ε, μου με τον Μοχάμεντ Ραμαντάν και τους οικείους του. Είναι ευθύνη όλων των ε, συνειδητοποιημένων πολιτών να αντιστέκονται στι αυθαίρετε συλλήψει, στα βασανιστήρια και τη θανατική ποινή όπου και αν συμβαίνουν. Επίσης, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να μιλήσω για την αδικαιολόγητη σύλληψη και κακομεταχείριση παιδιών. 237 παιδιά κρατούνται από τις αρχές του Μπαχρέιν, αυτές οι συλλήψεις μόνο το 2015. Πολλά εφίστανται κακομεταχείριση, ομολογούν εγκλήματα που δεν έχουν διαπράξει. Έχουμε παραδείγματος χάρη τον Σαΐντ Αλία Μπάς Μοχάμετ, τους αδερφούς Μοχάμετ Χασάν, και τον Σαΐντ Φεχέλ, τον Σαΐντ Σάμς και τον Σαΐντ Μοχάμετ Χασαμ. Όλοι έφηβοι που συνελήφθησαν τους τελευταίους μήνες και θα πρέπει να γυρίσουν στις οικογένειές τους. Το 2013 περάσαμε ένα ψήφισμα και ζητούσαμε από το Μπαχρέιν να σεβαστεί την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην οποία είναι συμβαλόμενο μέρος οι αρχέ του Μπαχρέιν πρέπει να απελευθερώσουν τον Μοχάμεντ Ραμαντάν και όλους τους ανήλικου κρατούμενου. Σας ευχαριστώ για τη διαδικασία και the Δύο λεπτά ο καθομιλητής, πρώτος ο κύριος Βόμποντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή πολλές είναι οι χώρες που αναζητούν τη σωστή εξισορρόπηση μεταξύ ασφάλεια και ελευθερία. Το Μπαχρέιν βρίσκεται στο σωστό δρόμο, όντω. Όμω δεν θα πρέπει να κοφεύουμε σε περιπτώσει όπω ε, η υπόθεση του Μουχάμετ Ραμαντάν και άλλων που περιμένουν να θανατωθούν. Θα μπορούσε να υπάρξει άφεση μόνο από τον ε, χάρη, μάλλον μόνο από τον αρχηγό του κράτους το, ή έστω μία ανάκληση της άσκησης θανατικής καταδίκης. Θα καλέσω λοιπόν τις αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειες μεταρρύθμισης της λειτουργίας των δικαστικών και αστυνομικών αρχών στη χώρα για να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η οπισθοχώρηση του Μπαχρέιν με την άσκηση της θανατικής ποινής και ο μη σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ένα φαινόμενο που έφερε σε πολλές περιπτώσεις συλλήψεων την άσκηση βασανιστήριων κατά την ανάκριση των ανθρώπων αυτών σε μεγάλη μάλιστα κλίμακα και παρά τις υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις. Στις 14 Φεβρουαρίου 2014 ο Αλή Μόζα και ο Ραμαντάν καταδικάστηκαν σε θάνατο από ποινικό δικαστήριο του Μπαχρέιν και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για τις αρχές, ε, μπροστά στην εισαγγελέα ομολόγησαν ότι παραδέχτηκαν ότι οι ομολογίες τους αποσπάστηκαν με την άσκηση βασανιστήριων. Η θανατική λοιπόν ποινή πρέπει να ανασταλεί και θα πρέπει να γίνει έρευνα ενδελεχής για την περίπτωση άσκησης βασανιστήριων των δύο αυτών ανθρώπων. Και η θανατική τους ποινή βεβαίως να ανακληθεί. Ευχαριστούμε Επίτροπος Κρετσού. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρε, εξαιρετικοί βουλευτέ, από το 2011 και μετά παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στον Μπαχρέν. Συστηματικά έχουμε επαφέ με τι τοπικέ αρχέ σε όλα τα επίπεδα. Σε διαρκή επαφή είμαστε με, με ένα ευρύ φάσμα ακτιβιστών και μη καπαόμικρων υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Παχρέν. Είναι σημαντικό εταίρο μα ε, στην περιοχή του κόλπου και είναι σημαντικό ο ρόλο του για τη σταθερότητα σε αυτή την περιοχή. Ο καλύτερο τρόπο για να επιτύχουμε τη σταθερότητα είναι να ενισχύσουμε το υφιστάμενο πλαίσιο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσωπικών ελευθεριών. Συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, τον, ε, ένα δραστήριο διάλογο, ένα ενεργό διάλογο με τις αρχές του Μπαχρέιν για όλα αυτά τα ζητήματα και πιστεύουμε ότι μετά την εθνική συμφιλίωση, η οποία οδηγεί σε μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, μπορούμε να βασιστούμε στην ανεξιθρησκεία και στο διάλογο για να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της περιοχής. Ε, φυσικά, όπως όλοι, ανησυχούμε και εμείς για θανατική ποινή, για τον Αλιμούσα και τον Ραμαντάν ε, και ε, μετά τη, που για το, τη βόμβα, το, την τρομοβιστική επίθεση του Φεβρουαρίου το 2014 όπου πέθανε ένας αστυνομικό και το 2015 εξεδόθηκε απόφαση από τον Άριο Πάγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά είναι κάθετα κατά τη επιβολή θανατικής επιγενής, όποιε και αν είναι οι περιστάσει, και είναι, παραμέ, θα, και θα παραμείνει ακρογωνίω λίθο τη εξωτερική μα πολιτική η απόρριψη της θανατική θανατικής ποινής. Φυσικά θα πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά αυτέ οι υποθέσει και στι Βρυξέλλες αλλά και ε, στην ε, επιτόπου αντιπροσωπεία μας ε, τόσο στο Ριάντ όσο και στον Μπαχρέιν ε, θα ε, συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές για να βοηθήσουμε τον Μπαχρέιν να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Υπάρχει και η ανεξάρτητη ερευνητική επιτροπή και έχουν εκδοθεί και συστάσεις στα πλαίσια της ε, διαδικασίας καθολικής αναθεώρησης του προγράμματος δράσης για τον Μπαχρέιν. Σε όλες τις περιπτώσεις σε, σε όλες αυτές τις ε, καταδίκες έχουμε προτείνει ε, προστασία των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Η τελευταία φορά ήταν το ΜΕΤΟ 2015 με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά είναι απάνθρωπη ε, αυτή η συμπεριφορά και την καταδικάζουμε περίφραστα σε όλες ε, τις ευκαιρίες ε, που έχουμε. Στη Μανάμα ε, στο Μπαχρέιν η αντιπροσωπεία μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και ε, παρακολουθεί γενικότερα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσημα πάρα πολλές φορές ε, έχει εκφράσει την άποψη ότι δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η χρήση βίας και επανειλημμένα ζητά διαφανείς διαδικασίες διερεύνησης όλων των υποθέσεων ε, αδικαιολόγητων ε, βασανιστήριων ε, και με διαφανή τρόπο θα πρέπει να λειτουργεί το Μπαχρέιν όπως προκύπτει και από τις συστάσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής του Μπαχρέιν και να δρά για το κοινό καλό. Έχουν ε, αναλυθεί ήδη πολλά μέτρα από τις αρχές του Μπαχρέν για την εφαρμογή των συστάσεων της ανεξάρτητης ε, εξεταστικής επιτροπής. Είναι σημαντικά αυτά τα βήματα και αναβαθμίζουν την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν επαρκούν όμως ο διαμεσολαβητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων και η Διεθνής Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν ε, εκπληρώνοντας την την εντολή τους ε, με πλήρη διαφάνεια και ε, ανεξαρτησία. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω και πάλι για το ότι θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε τις δύο περιπτώσεις αυτές, ε, Αλιμούσα και ραμαντάνε και από τους ενδειγμένους διάβλους επικοινωνίας θα συνεχίσουμε να δρούμε. Ευχαριστούμε. Συνάλφοι, 7 προτάσεις ψηφίσματος.